Βάζω την ικανοποίησή μου που ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία που θα βελτιώσει την διακίνηση μεταξύ Ευρώπης και Βιετνάμ. Πέρα τη συζήτηση θα ψηφίσουμε σήμερα στις 11.30. Τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Μπαλτζάνη για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012. Αφήνω τον Επίτροπο να καθίσει και δίνω το λόγο στην κυρία Μπαλτζάνη για τέσσερα λεπτά. Το έγγραφο το οποίο εξετάζουμε σήμερα δεν είναι μόνο ένα έγγραφο για τις προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού, Πρόκειται κυρίως για ένα στρατηγικό έγγραφο για το νέο ρόλο που θα πρέπει να αποκτήσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Πρόκειται για, φέτος για ένα ευρωπαϊκό στην κυριολεξία εξάμεινο για την εναρμόνιση και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικού και εθνικών προϋπολογισμών. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει σύγκληση. Σύγκληση των προϋπολογισμών των κρατών μελών προς τους μεγάλους ε, στόχους ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι ευρωπαϊκή στόχοι σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλοι από αυτούς της Ευρώπης 2020. Μια μεγάλη στρατηγική φιλόδοξη με πέντε βασικούς στόχους. Μεγάλη στόχη, αλλά και ιδιάζονται στόχοι. Πρώτο, μία καλύτερη Ευρώπη, καλύτερα απασχολούμενη Ευρώπη μέσα από μεγάλες επενδύσεις. Για το 2012 έχουμε μεγάλους στόχους, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο πρώτος στόχος, περισσότερη εργασία στην Ευρώπη. Είναι θεμελιώδες και επίγον να ορίσουμε ευθύ αμέσω τη διάσταση της στρατηγικής του 2020 στον προπολογισμό μας. Χρειάζονται δύο θεμελιώδη πράγματα. Πρέπει να σχεδιάσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Να αποκλείσουμε μαθηματικές εφαρμογές στον προπολογισμό δεν έχει νόημα. Η μαθηματική εφαρμογή δεν είναι χρήσιμη πρέπει να δούμε ποια είναι τα χρήσιμα προγράμματα και οι χρήσιμες δράσεις για τη στρατηγική μας του 2020. Και το να ταινίζουμε το μέλλον σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, διότι με τις δεσμεύσεις οικοδομούμε εμείς το αηφόρο μέλλον της Ένωσης, όχι με τις πληρωμές. Και υπάρχει και το θέμα της ευκαμψίας ολοκληρώνουμε τη φάση προγραμματισμού. Και ο προϋπολογισμός είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να δούμε όλα τα μέσα ευελιξίας που έχουμε ως θεμελιώδη και παραβάτως απαραίτητα για τον προϋπολογισμό μας σήμερα. Αυτό είναι ουσιαστικότατο για να καταλήξουμε στη στρατηγική του 2020 που δεν πρέπει να πτωχεύσει. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχουμε ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν με υπονομή από κοινού ξεκινήσουμε ένα ανανεωμένο κλίμα διαθεσμικής συνεργασίας που πρόκειται για μία από τις τεράστιες προκλήσεις της Λισαβόνας. Δεν μιλάμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα. Χρειάζεται μία ανανεωμένη ισοτομία για να ισοτιμία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στον προϋπολογισμό στρατηγικά για την οικοδόμηση του μέλλοντος. Ο κύριος Λεβαντόφσκι εξ ονόματος της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Μπαρτζάνη. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λεβαντόφσκι, για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι όπως ε, αντικατοπτρίζεται στην έκθεση βάσει των κατευθυντηρίων μας γραμμών. Η Επιτροπή που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας φυσικά και πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από την άλλη μεριά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πιο πρόσφατα στοιχεία που μας έρχονται από τις 27 χώρες μέλη. Τα ελέγχουμε λοιπόν, τα αξιολογούν οι υπηρεσίες μας προκειμένου να ε, δώσουμε μορφή στη συνέχεια και στις αποφάσεις που θα ληφθούν στις 20 Απριλίου. Τώρα είμαστε στη δεύτερη δοκιμασία της ετήσιας διαδικασίας βάσει της ηθικής της Λισαβόνας. Το πλαίσιο είναι σαφές για όλους. Είναι ένα πλαίσιο οικονομικής σταθερότητας. Πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι λοιπόν σημαντικό να ανταποκριθούμε σε όλε τις δημοσιονομικές υποχρεώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά όμως αυτό να το κάνουμε στα πλαίσια μιας λιτότητα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η προσπάθεια να ετοιμαστεί ο προϋπολογισμός σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό αυτό. Και είναι σημαντικό επίσης να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε την Ευρώπη σήμερα που βρίσκεται στην περίοδο μετά την κρίση. Και θέλω να σας θυμίσω δύο διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους εθνικούς προπολογισμού και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικοί αναφέρονται ε, στα κοινωνικά δικαιώματα, στην κατανάλωση, στις δαπάνες. Ο ευρωπαϊκός ε, προπολογισμό όμως πρέπει να φροντίσει για την ανάπτυξη δεν είναι δυνατόν βέβαια να μην τηρήσει τις υποχρώσεις που έχει αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε προκειμένου να ετοιμάσουμε τον προπολογισμό για το 2012. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας το έχει πει και το λέει και στην έκθεσή της η κυρία Παντσάνη, Πρέπει να φροντίσουμε για αρκετή χρηματοδότηση όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής μας 2020 Όντω πρέπει να το κάνουμε αυτό. Συγχρόνω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται για τις διοικητικέ μας δαπάνες. Και γι' αυτό έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δαπανίσει να δώσει λιγότερο από 1% αύξηση όσον αφορά τις διοικητικές της δαπάνες και να φροντίσει να υπάρχουν και εξοικονομήσεις για τις διασκέψεις, τις αποστολές, ε, τεχνολογία κλπ λαμβάνοντας υπόψη τόσα έγιναν πέρυσι, λαμβάνοντα υπόψη την εμπειρία που έχουμε από την ετήσια διαδικασία προετοιμασίας του προπολογισμού για το 2011, πιστεύουμε ότι φέτος θα προχωρήσουμε πιο εύκολα. Προσδοκώ την πρώτη μας συνάντηση, τον τριμερή διάλογο στις 30 Μαρτίου και μετά θα ετοιμάσουμε και το σχέδιο προπολογισμού μας για το 2012. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Τώρα εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Λάβια για δύο λεπτά εκ μέρου του Αξιότιμοι Πρόεδρε, αξιότιμοι Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Το ΕΛΚ για τον προϋπολογισμό του 2012 απ' την αρχή υποστήριξε την δημιουργία ενός ιεραρχημένου σχεδίου προτεραιοτήτων για να το παρουσιάσει στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Εμείς συμβάλαμε στο να διευρύνουμε το σπέκτρο των κοινοτικών πολιτικών και συμμεριζόμαστε την ισορροπημένη θέση της εισηγήτριας όπου εισήγαγε την ανάπτυξη και την έρευνα και την καινοτομία ως προτεραιότητες που είναι προτεραιότητες που συμμερίζεται από πάντα το ΕΛΚ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα πρέπει να μας παρουσιάσει η Κομισιόν. Η ευθύνη θα πρέπει να αποτελεί, όπως είπε και ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι, το κύριο χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού 2012. Αλλά σήμερα, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω της κρίσης, πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές από τις χώρες της Βορείου Αφρικής και για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την, το να μπορέσουμε το να μην μπορούμε μάλλον να παρεύουμε όταν συμβαίνουν απρόοπτα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό όμως πρέπει να σας πω ότι η πρόταση της ΓΚΟΕ για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν έχει κανένα νόημα. Είναι κάτι το εντελώς ασήμαντο. Ο κύριος Φέρμου για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ε, η συγγήτρια είναι πολύ καλό σημείο ε, κίνησης για την έκθεση του. Σύντομο, επικοδομητικό και τονίζει τα πιο σημαντικά θέματα. Ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά θέματα. Είναι να καταδεχθεί ότι η στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο κενό γράμμα, αλλά είναι μια πραγματική προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Πρόκειται μόνο για ένα μικρό τμήμα του συνολικού κόστους, αλλά μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο όταν πρόκειται για την επένδυση σε σχέδια τα οποία δεν μπορούν να υπομισθούν από μόνα τους κάποια κράτη-μέλη ή που απαιτούν αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Έρευνα και ανάπτυξη, υποδομή για την τεχνολογία και τις μεταφορές, εφαρμογή δηλαδή πραγματική της εσωτερικής αγοράς και ανάπτυξης του πλήρους δυναμικού Μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά για να μπορέσει έτσι να ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια κοστίζουν χρήματα και γι' αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί από πλευράς κρατών μερών και συμβουλίου ότι πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Αν θέλουμε να λειτουργήσει το σύστημα 2020 ε, πρέπει να γίνει αυτό. Αλλιώ, όπω η στρατηγική τη Λισαβόνα θα εξακολουθεί να παραμένει καινογράμμα. Ευχαριστώ, κύριο Σάκλου. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εισαγωγικά θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μα. Τη σήμερα ημέρα δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανεί δημοσιονομικέ προτεραιότητε. Οι στόχοι της Ευρώπης 2020 είναι πολύ σημαντικοί βέβαια. Δημοσιονομικά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο το 2014 δηλαδή για να καθορίσουμε τον προπολογισμό μας όσον αφορά τους στόχους του 2020. Η Επιτροπή λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη της την επόμενη πρόταση για τον προπολογισμό και τους στόχους αυτούς, πράγμα το οποίο σήμερα δεν έχει γίνει ε, μέχρι τώρα. Όπως είπε και ο κύριος Φάρμ, πρέπει να φροντίσουμε οι στόχοι αυτοί να γίνουν πραγματικότητα και να μην καταλήξουν στο σιρτάρι ενός γραφείου. Η ομάδα μου έχει καταθέσει διάφορες τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Και χαιρόμαστε γιατί έχουν συμπεριληφθεί τώρα στην έκθεση από την εισηγήτρια, πράγμα για το οποίο θέλω και να την ευχαριστήσω. Στο Συμβούλιο πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στο Κοινοβούλιο πρέπει εμείς να έχουμε ένα μορατόριο και να δούμε τι θα κάνουμε με τον προπολογισμό του 2011. Έτσι κι αλλιώς υπήρξαν διαμάχες ε, και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ξέρουν αυτό όλοι οι πολιτικοί. Έχουμε όμως λόγο να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, με κάποιες οικονομίες στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νέε εξουσίε σήμερα και το Συμβούλιο έχει την εντύπωση ότι αυτές οι νέες αρμοδιότητες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας τις δημοσιονομικές. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και θέλουμε μια επικοδομητική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουμε καλέ διαπραγματεύσει όσον αφορά τον επόμενο προπολογισμό. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Έλλη έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για την έκθεσή τη. Άλλες κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε συζητήσει ε, εδώ τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Αυτή τη φορά υπάρχουν ε, περισσότερες λεπτομέρειες, είναι καλύτερες. Η ομάδα μου πάντως πιστεύει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην περιοριζόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες. Η παράγραφος που θέλουμε εμείς για την παράγραφο 21, εκεί που λέμε για τις ε, εξοικονομήσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όντω πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες. Μέχρι τώρα έχουν γίνει ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η επιθυμία να έχουμε χρήματα για να διατύχουμε τους στόχους της Ευρώπης του 2020. Όντως, αλλά ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και αλλιώς, όχι μόνο οικονομικά, δεν πρόκειται μόνο για χρήματα, μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, να έχουμε και άλλες δράσεις ώστε να μπορέσουμε συγχρόνως να εξοικονομήσουμε από τον προϋπολογισμό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα πρέπει να σου πούμε θέλετε περισσότερα χρήματα, φροντίστε να τα εξοικονομήσετε από κάτι άλλο τότε. Έτσι θα προχωρήσουμε. Πρέπει να δούμε τι ευθύνες θα ε, αναλάβουμε εμείς για την λιτότητα δεν είναι δυνατόν να κάνουμε οικονομίες εκεί που πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα. Όχι, αλλά πρέπει να παγώσουμε τις δαπάνες μας γενικά για το 2012. Η κυρία Τρούπελ για τρία λεπτά τώρα. Κύριε Πρόεδρε, εξαιρετική κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Ναι, και εμεί οι πράσινοι θεωρούμε ότι στι εποχέ που δεν έχουμε πολλού δημοσιονομικού πόρου και υπάρχει δυνατότητα πολιτικής λιτότητας, πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν μειώσεις στα, κρατικό... στα αλλά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μπορούμε να χρεωθούμε ευτυχώ. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο μειώσει, αλλά εξέβρεση μια ισορροπία, ούτω ώστε να επενδυθούν χρήματα σε σχέδια που πραγματικά προωθούν στο μέλλον για να μην διακυβευθεί η οικονομία. Αυτά πρέπει να είναι και η κατευθύνια γραμμή για τον προπολογισμό του 2012, αυτή η ισορροπία δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια αναλάβαμε στα πλαίσια των ελευθερωτικών ταμείων υποχρεώσει μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού που πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα επόμενα έτη. Θεωρώ ότι η προσέγγιση της κυρίας Μπαρζάνη να πάρει δηλαδή τα κεντρικά σημεία της στρατηγικής του 2020 για να δει προς τα που θα κινηθούμε είναι πάρα πολύ καλή. Ε, κλιματικές αλλαγές παραδείγματος χάνει. Πιο γλίγορα είσοδος στις ανασυνώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότεροι πόροι για την παιδεία και την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι στόχοι που θα πρέπει να τηρήσουμε, δεν θα πρέπει να τους διακυβώγουμε. Θεωρώ επίσης σωστό ότι με το μέσο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καταβάλλω τώρα προσπάθειες ούτως ώστε τα κράτη-μέλη με τους προπολογισμού τους και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 28 προπολογισμοί δηλαδή θα πρέπει να προωθούν τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Πού θα πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα. Εάν δούμε τώρα την δημοκρατική αλλαγή ελπίζουμε στις αραβικές χώρες βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εκεί περισσότερη ε, <clears throat> κοινωνία των πολιτών, δημοκρατία και πρέπει να τους υποστηρίξουμε στον δρόμο τους αυτό προς μια δημοκρατία. Χρειαζόμαστε περισσότερους σπόρους για να προωθήσουμε τη δημοκρατία στον κόσμο. Σπράσινοι βουλευτή, θέλω να σας πω και εν ώψη της Ιαπωνίας και πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Πιστεύουν οι πράσινοι μπορούμε να εξοικονομήσουμε στον ε, αντιδραστήρα και την πυρηνική σύνδεξη ΣΥΤΑ. Γιατί χρειαζόμαστε τόσα χρήματα για να ξεκινήσουμε το σχέδιο αυτό αντί να μεταχειριστούμε τους σπόρους σε βρατό για να βγούμε από την πυρηνική ενέργεια και να μπούμε πολύ πιο γλύτερα σε ανενώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε όλοι αν έχουμε κατά νου τον ΟΗΕ και την ε, πολιτική κλίματος ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη μορφή ε, ενέργειας που παράγουμε. Και ο προεπολισμός 2020 Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβάλλει προς τα αυτά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με τις νέες δημοσιονομικές προβλέψεις να πραγματοποιήσουμε αυτού του τύπου τις ποιοτικέ αλλαγές. Ευχαριστώ κύριε Τρίπελη Πρόεδρος. Ο κύριος Πόρτας, μισή λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ενώ εμείς εδώ συζητάμε τους προσανατολισμούς το 2012, απ' έξω δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων μας στέλνουν ένα σαφέστατο μήνυμα μας λένε ότι η πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη πνίγει την οικονομία και βλάπτει τις συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων. Λένε αυτοί οι πολίτες το ευρωπαϊκό μοντέλο, το, το οικονομικό συγγνώμη, μοντέλο το οποίο επιβάλλεται δεν εγγυάται σε τίποτα την αηφόρο ανάπτυξη και την δημιουργία απασχόλησης. Μας λένε ότι το σύμφωνο για το ευρώ το οποίο θα εγκρίνει σήμερα η διάσκεψη κορυφής είναι ένα σύμφωνο το οποίο θα βλάψει τις αγορές και τον κοσμάκι που θα πληρώσει για μια κρίση που δεν δημιούργησε ο ίδιος. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της διαμαρτυρίας. Θέτει κάτι το ουσιαστικό στην όλη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ποιες είναι οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Μας λένε οι συντηρητικοί θέλουμε έναν προϋπολογισμό με μηδενική αύξηση. Ακούσαμε και άλλους να λένε ότι λόγω της πολιτικής λιτότητας θα πρέπει να έχουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με μία αύξηση μηδέν. Αυτή είναι η λάθος απάντηση και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση για έναν απλό λόγο. Δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε πολιτικές λιτότητες σε εθνικό επίπεδο πάντα πιο ισχυρές και μετά να λέμε ότι λόγω των πολιτικών λιτότητας χρειαζόμαστε πάντα έναν μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με ένα τέτοιο σκεπτικό εμείς καταλήγουμε στην, σε, βασικές επιπτώσεις λιγότερες δημόσιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη κοινωνική παρακμή. Αυτή είναι η βασική προβληματική του προϋπολογισμού του 2012. Θα πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό που να μειώνει τις ανιτότητες. Αυτή η έκθεση είναι γεμάτη από καλές προθέσεις αλλά δεν απαντάει σαφώς στην πρόκληση που μας θέτει ο κόσμο της εργασίας. Η κυρία εν δύο λεπτά. Μια δυναμία είναι το να ξεχνάμε τις παρατηρήσεις που έχει κάνει το Ελεκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του. Εμείς πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι η μόνη διαθέσιμη πληροφορία μιλάει για αποτελεσματικότητα. Ότι αποτελεσματικότητα πρέπει να υπάρχει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να θέλουμε να αυξάνουμε τον προπολογισμό για να ανταποκριθούμε στην ε, στρατηγική του 2020 πιστεύοντα ότι έτσι θα βγούμε από την κρίση, μα κάνει να ξεχνάμε την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Υπάρχει απειλή ότι περιορίζοντας τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσφέρουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το ρυθμό των, της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο μας ε, οδηγεί να αγνοούμε τελικά την κατάσταση που επικρατεί ακριβώς εκεί. Ως ε, φορολογούμενοι ζητάω και από τον Κάμερον να φροντίσει για μια προσαρμογή του προπολογισμού του 2012. Έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουν αυτά που θέλω εγώ. Η κυρία Βέτμα τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις σημεία της ε, κυρία της κυρίας Βολσάνη. Καταρχήν η έκθεση για το προπολογισμό 2012 ε, βασίζεται στην προϋπόθεση του καλύτερου διακανονισμού της ευρωπαϊκής ε, και οικονομικής πολιτικής του, του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Επίσης, κάτω από τις κατευθύνσεις γραμμές της πολιτικής για το 2020, η βελτίωση του επίπεδου παιδείας και η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, που είναι για μένα τα βασικά σημεία για την δυνατότητα λειτουργία της Ευρώπης. Δεύτερον, τονίζει την αναγκαιότητα βελτίωσης της συνεργασίας ε, των επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι. Καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συμφωνία και συγκέντρωση σε λογικούς πόρους, ε, στόχους, συγγνώμη, είναι πράγματα που θα πρέπει να υποστηρίξουμε για να βελτιώσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Τρίτον, ε, στόχοι ενέργειας και κλίματος. Εν ώψη της καταστροφής στην Ιαπωνία θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δημιουργία οικολογικών θέσεων απασχόλησης δεν θα οδηγήσει μόνο στην επίτευξη των κλιματολογικών στόχων, αλλά είναι πολύ σημαντικές και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να ε, παρουσιάσει χρέος. Και γι' αυτό ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μόνο το 2% των δημοσίων δαπανών εδώ. Ευχαριστώ. Εξονόμητος των άλλων ομιλητών. Καταρχήν ο κύριος Γαρίδα Πολέδο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να αρχίσω ξεκινώντας, ευχαριστώντας την κυρία Μπαρσάνη για την ευελιξία της, διότι η αρχική ιδέα δεν πρόβλεπε να συζητήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, πράγμα όμως που αποδείχτηκε πολύ θετικό για τη λιτότητα. Η λιτότητα δεν είναι μία αρχή, είναι ένα μέσο. Ένα μέσο για να καταφέρουμε κάτι, για να καταλήξουμε σε έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό και που να μην μας οδηγεί αυτό το οποίο εκεί που οδήγησε η πραγματικότητα σε πολλές χώρες δημιουργώντας εξωπραγματικές καταστάσεις και πολιτικά προβλήματα. Δεν θα πρέπει στην ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού να εντάσσουμε ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο, σε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ο φόρος ε, για την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών πράξεων εντάσσεται σε ένα πολυετές πρόγραμμα. Το να εντάσσουμε αυτή τη συζήτηση σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό μπορεί να μας οδηγήσει σε μία λάθος διαπραγμάτευση, ε, σε μία λάθος στρατηγική διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να βάζουμε σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό ιδέες ή μέτρα τα οποία εντάσσονται σε ένα πολιετές πλαίσιο. Για να μην καταλήγουμε όπως εμείς το 2011 με ένα περιθώριο πιστώσεων πληρωμών που ξέρει πολύ καλά ο κύριος Επίτροπος δεν μας επιτρέπουν να πληρώσουμε και τις βραχυπρόθεσμες πληρωμές. Ευχαριστώ κύριε Γκαϊέρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κυρίε και κύριοι, συζητάμε σήμερα την αναγκαιότητα να κάνουμε εξοικονομήσει εν ώψη μιας ε, κρίση χρέους που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. του ε, Τρουπέλ Δικαίω αναφέρθηκε όπως και άλλοι στην κρίση αυτή και που μας πλήττει μόνο έμεσα γιατί εμείς στον κοινοτικό προπλησμό δεν επιτρέπεται να αναλάβουμε χρέος. Τι θα μπορεί να γίνει όμως εάν το 2% των δημοσίων δαπανών των 27 κρατών μελών είναι μονάχα ο προβλεπισμός της Ένωσης. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μία πολιτική λιτότητα αλλά να θέσουμε κάποια σύμβολα. Σύμβολα που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη, δίνουν την εντύπωση ότι τα κρίματα που αποστείλουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίζονται, χάνονται. Θα πρέπει όμως να μην ε, ξεχνάμε ότι πρέπει να παρουσιάσουμε ότι οι πόροι αυτοί επανέλθονται στα κράτη-μέλη, όχι ένα προς ένα βέβαια, γιατί δεν είναι ταμιευτήριο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ακολουθεί και μια πολιτική αλληλεγγύης υποστηρίζοντας εκείνες χώρες που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες. Αλλά το κάνει στην Βόρεια Ρινανία ε, στη χώρα μου πολλά σχέδια ε, συγχρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν αυτά τα χρήματα σταματούσαν θα χάναμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Στην ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου λέω ότι τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για τις δαπάνες, στις των ευρωπαϊκών χρημάτων δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Διαβάζω επίσης ότι η επανάκτηση, η επιστροφή των ε, χρημάτων αυτών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως είναι δισεκατομμύρια. Και βλέπω ότι εκεί που δεν υπάρχει σωστή διαχείριση ε, των κοινοτικών χρημάτων πρέπει να σταματήσει όπως γίνεται στη Γερμανία ή στον, ε, στην ελλαδα Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η χρηματοδοτηση ευρωπαικη ενωση θα πρεπει χρήση των χρημάτων αυτών, να βελτιωθεί η διαχείριση, πράγμα που θα μας επιτρέψει να δαπανούμε καλύτερα τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Όχι περισσότερα, καλύτερα λέω. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γέντσεν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μπαρσάνη. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά μας, αλλά πολύ δύσκολο το έργο μας για να ετοιμάσουμε τον προπολογισμό αυτό. Και αυτό γιατί το πλαίσιο είναι δύσκολο. Ο προπολογισμό είναι έτσι που έχουμε περιορισμούς όλο και περισσότερους με τις δημοσιονομικές προπτικές. Για παράδειγμα, οι αγροτικές δαπάνες χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτηθούν νέες πρωτοβουλίες, επενδύσεις, για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας. Η Άρα είναι όλο και πιο δύσκολο να υπάρχει πραγματική συνοχή στις δαπάνες. Συμφωνώ με τους πράσινους πάντως που λένε ότι δεν πρέπει να δώσουμε χρήματα για το ίτερ, για την πυρηνική σύνδεξη Πρέπει να θυμόμαστε τι συνέβη στην Ιαπωνία. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και, υπάρχει και το θέμα των στερεών καυσίμων. Το 2012 πρέπει να βρούμε άλλα μέσα. Και χαίρομαι που ο Επίτροπος μας λέει ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ίδιος όπως και εκείνος των χωρών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον πρέπει να πληρώνει τους λογαριασμούς της. Ο Επίτροπος θέλει να έχουμε πιο εύκολες διαπραγματεύσεις αυτή τη φορά και έτσι πιστεύει ότι θα πάνε πιο εύκολα οι διαπραγματεύσεις. Όντω και εμεί από τη δικιά μα ε, την πλευρά πρέπει να κάνουμε πιο συγκεκριμένε προτάσει, λαμβάνοντα υπόψη τι πραγματικέ ανάγκε. Τέλο, ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που επέμεινε για το ότι πρέπει να γίνουν ε, οικονομίες στις διοικητικές δαπάνες. Είναι μία από τις θέσεις όπου πράγματι μπορούμε να πετύχουμε οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της αυτή την ε, πλευρά και θα γίνει το ίδιο και στα άλλα θεσμικά όργανα, όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Φάντμον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε και κύριοι. Ο προπολισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 θα πρέπει να ε, ακολουθήσει την παράδοση ισορροπημένου προϋπολογισμού Δεν πρέπει να περάσουμε στις διαφωνίες που είχαμε το 2011. Δεν επιτρέπεται να έχουμε ένα προσωρινό προϋπολογισμό πάλι, γιατί αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφύγουμε τις διαφωνίες αυτές και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τον γρηγορότερο τον, τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε καλή πρόταση προϋπολογισμού, πάντα που σημαίνει σήμερα η να κάνουμε οικονομίες. στα κράτη-μέλη περιμένουν σε εποχές λιτότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, φέρεται όπως πρέπει στον τομέα αυτό. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα αξιοπιστίας. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό κύριο Σφερέρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει εναλλακτική λύση στη συνένεση μεταξύ της δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Συνένεση η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά και σίγουρα όχι στην έξοδο από την κρίση. Η εναλλακτική λύση σημαίνει τι, σημαίνει μια βαθιά μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε μια φάση που εντείνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και ο κοινοτικός προπολογισμός θα πρέπει να μας οδηγήσει σε πραγματική σύγκληση, θα πρέπει να οδηγήσει στην αξιοποίηση ε, των κοινωνικών δυνάμεων όλων των χωρών θα πρέπει να, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης στην εγκρίζωση της φτώχειας θα πρέπει να αποτελεί ένα μοχλό εξόδου από τις κρίσεις. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε την... τον δρόμο που προβλέπει η στρατηγική του 2020 και που θα οδηγήσει σε μία αύξηση των περιφερειακών και κρατικών ανισοτήτων. Θέλουμε μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αλληλεγγύη και για την αηφορία που να βασίζεται σε νέες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που θα υποστηρίζονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και αυτό το έχουμε καταγράψει με αλλαγές στις διάφορες, στην έκθεση. Θα πρέπει ο προϋπολογισμός να αποτελεί επίσης ένα μοχλό ειρήνης και όχι έναν, ένα μέσο διάδοσης πολέμου και επεμβάσεων. Θέλουμε ένα νέο δρόμο για την Ευρώπη. Ο κύριος Μοργάντη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι νέοι προσανατολισμοί του προϋπολογισμού θεωρώ ότι είναι κενή νοήματος δεν ορίζονται οι πραγματικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για την κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού. Αναφέρεται συχνά η στρατηγική του 2020. Πρόκειται όμως για μια μεγάλη και δαπανηρή στρατηγική. Ποιες θέλουμε να είναι οι προτεραιότητες μέσα σε αυτήν τη στρατηγική του 2020. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους ήδη κουτσουρεμένους ε, προϋπολογισμούς ε, και να εκτιμήσουν το τι θα πρέπει να κάνουν και να ορίσουν τις προτεραιότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας αυτοσκοπός. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν ορίζει τίποτα καινούριο. Ο κύριος Χάρτον, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ η, από τη Σοσιαλιστική Ομάδα Βαρζάντη μας ετοίμασε αυτήν την έκθεση η οποία όμως προβλέπει ένα προπολογισμό όχι καλό για τους πολίτες, για τον εαυτό της. Λέει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σωστές σχέσεις και με τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάμε πόσα χρήματα έχουμε εξοδέψει. Για το Γαλιλαίο, για παράδειγμα. Για μένα είναι σαφές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα με μια τέτοια πρόταση. Χρειάζεται όμως υπευθυνότητα και βιωσιμότητα. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σαφής. Είναι νόητη η έκθεση αυτή. Δεν είναι αυτό που θέλουν και που προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχει καμία φιλοδοξία για εξοικονομήσεις. Αντίθετα μιλάει για σπατάλη ακόμα περισσότερου χρήματος. Δεν, η σοφία λένε ότι έρχεται με τα χρόνια. Δυστυχώς όμως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό δεν συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Σουριάν τώρα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα πρότεινα, αγαπητοί συνάδελφοι, να αφήσουμε τις φλιαρίες και να περάσουμε στην πραγματικότητα. Δεν ήταν εύκολο για την εισηγήτρια να προετοιμάσει αυτή την έκθεση, γιατί δεν μπορούμε ακόμα να σας μιλήσουμε για αριθμητικά στοιχεία, μια που η Κομισιόν δεν έχει ακόμα υποβάλει καμία πρόταση για το πλαίσιο του προπλογισμού. Για τις αρχές μπορούμε να συζητήσουμε μακρόν Και η εισηγήτρια έθεσε το θέμα πάρα πολύ σωστά. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να εντάσσουμε την στρατηγική του 2020 στο πλαίσιο του προπολογισμού. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουν τεθεί ακόμα πλαίσια για τις επιμέρους πολιτικές ανατομέα και δεν αναφέρονται καν οι πολιτικές αυτές, μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες κριτικές παρατηρήσεις γιατί χωρίς αυτούς τους στόχους το θέμα είναι πολύ αόριστο θα έλεγα. Αυτό που μπορούμε να, συμφωνήσουμε είναι ότι η πολιτική συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αυτή τώρα ξεκινάει να αναπτύσσεται και να βοηθά στην ανάπτυξη. Εν αντιθέσει ε, από πολλούς που, άλλους που πήραν τον λόγο, θέλω να τονίσω ότι οι πληρωμές αυτές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν πρόκειται για σπατάλη χρημάτων, αλλά πρόκειται για δαπάνες που προωθούν την Ευρώπη, γιατί ακριβώς οι μειονεκτούσες περιοχές παίρνουν κάποιους πόρους και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ζητήσει το Κοινοβούλιο, να φτάσουν δηλαδή οι επενδύσεις εκεί που χρειάζονται. Αυτού του τύπου οι επενδύσεις, όχι οι επενδύσεις ε, ε πολυτελείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κρελικ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Μπαλτσάνη για την συνεκτικότητα των προτάσεών της ε, για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού. Στέλνει ένα σαφές ε, μήνυμα ένα σαφές πολιτικό μήνυμα στο ύψος των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων της στιγμής, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας πιο μακρόπνοης στρατηγικής. Εμείς ε, σήμερα θα πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τους διαδηλωτές ε, των Βρυξελών ε, για να απορρίψουμε αυτές τις αμφισβητήσιμες οικονομικές πολιτικές οι οποίες οδηγούν στη διαμόρφωση διαρθρωτικής ανεργίας στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά ορίζεται σαφώς ο νέος προϋπολογισμός του 2012 ατενίζοντας τις γραμμές του, της Ευρώπης 2020. Χρειάζονται προτεραιότητες, προτεραιότητες γιατί η στρατηγική 2020 ορίζει απασχόληση της τάξεως του 65%. Ο κύριος Λεβαντόφσκι βέβαια δήλωσε <coughs> στο γαλλικό τύπο πριν ρωτήσει το κοινοβούλιο ε, δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν αποφασίσει την απόλυτη λιτότητα και τη θεωρεί συμπληρωματικό κόστος όχι σύμμαχο φιλόδοξων πολιτικών. Η διαδικασία του προϋπολογισμού θα αποτελ... του 2012 δεν θα μπορέσει να είναι μια μακρόπνοη πολιτική εκφράζοντας μόνο το 2% των εθνικών ευρωπαϊκών προϋπολογισμών. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε πολιτικές, θα απομονώσουμε τους πολίτες αντί να τους προσετεριστούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπε για την ανακοίνωσή σας για τους ίδιους πόρους. Ευχαριστώ. Όταν χτίζει κανεί ένα σπίτι, συνήθω τον βαρύ λογαριασμό τον παίρνει στο τέλο. Στην αρχή συμφωνεί με τα έξοδα. Ε, το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Δηλαδή, στο τέλος έρχεται ο μεγάλο λογαριασμός, που δεν το ξέρουμε από πριν. Προσοχή λοιπόν τι πληρώνουμε και προσοχή τι κάνουν διάφορες χώρες, όπως η Ολλανδία, η οποία τελικά έχει μια κυβέρνηση την οποία δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Συμφωνούμε με την προσφορά, και γι' αυτό τελικά πρέπει να πληρώσουμε και ολόκληρο το λογαριασμό. Όταν στο τέλο τη διαδικασία προσπαθεί να εξοικονομήσει χρήματα και να κάνει οικονομίε, βέβαια δεν γίνεται και σωστά το λέει αυτό και η συγκήτρια. Αλλά όπω και να έχει το πράγμα θα πρέπει να πληρώσουμε τον τελικό λογαριασμό. Και το να αντιστεκόμαστε σε αυτό μας κάνει απλώς αναξιόπιστους και δημιουργεί και αισθήματα κατά της Ευρώπης στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κ. Λαμασούρ δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, τι να κάνουμε. Οπότε περνάμε στην κυρία Έρτσοκ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προπολογισμός 2012 είναι ο έκτος μέσα στα πλαίσια αυτών των δημοσιονομικών προβλέψεων και γι' αυτό ε, έχουμε τώρα πια μια σαφή εικόνα όσον αφορά τι ελλείψεις και τις θετικές εξελίξεις ε, ο προβλησμό του 2012 θα πρέπει να μα επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε τους στόχου και τι προτεραιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωση, ιδίως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής Ευρώπη 2020. Αυτό θα μας βοηθήσει να βγει πιο εύκολα η Ευρώπη από την κρίση, ιδίως πιο ενδυναμωμένη με έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη, ε, προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας, προώθηση της κοινωνικής ε, ολοκλήρωσης και καταπολέμηση της φτώχειας. Η στρατηγική του 2020 μπορεί να είναι μόνο αξιόπιστη αν μπορεί ικανοποιητικά να χρηματοδοτηθεί. Και εδώ θα ήθελα να υποθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο τόνισε πολλές φορές αυτές τις σημαντικές πολιτικές ε, επιφύλαξεις. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε να μην έχουμε λιγότερη Ευρώπη σε μια ε, παγκόσμια κατάσταση όπου υπάρχουν καταστροφές φυσικές και ανθρωπογενείς και καταστρέφουν τη ζωή πολλών. Αυτές δεν αφορούν μόνο μια χώρα, μια περιφέρεια, αλλά πολλές χώρες, όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και κοινωτικού πόρους για να πραγματοποιήσουμε στόχους μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμαϊερ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο προπολογισμό 2012 βρίσκεται ενώπιον δύσκολων εποχών για τα 27 κράτη-μέλη. Γι' αυτό δεν θα μπορούμε μάλλον να πληρώσουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να ε, χρηματοδοτήσουμε. Ε, θεωρώ ότι η έκθεση κ. Βασάνη είναι μια ανεκτή συμβαστική πρόταση. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες επικρίσεις γιατί περισσότερα χρήματα για μένα δεν σημαίνει αυτόματα περισσότερη ελληνική και περισσότερη Ευρώπη. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα των χρημάτων που δαπανούνται και ιδίω να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, να μην δαπανίσουμε απλώ τα χρήματα. Επίσης, ενδεχόμενοι είναι ήδη οι πόροι. Είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά γιατί θα πρέπει να οδηγήσει σε συμπληρωματική επιβάρηση των πολιτών ή των επιχειρήσεων που πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές παγκοσμίω. Θεωρώ επίσης σημαντικά να μην τονίζουμε συνέχεια ότι ο προβληματισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο το 2% γιατί πολλές χώρες χρηματοδοτούν πολλά ευρωπαϊκά σχέδια, άρα η επιβάρυνση για τις χώρες αυτές είναι μεγαλύτερη. Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό η έρευνα, η παιδεία και η βιώσιμη μορφή της οικονομικής ανάπτυξης να προωθηθούν και γι' αυτό μεγάλα σχέδια όπως η και ευχαριστώ την κυρία Γένδη για τις ε, παρατηρήσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ξεκάθαρα αλλιώς θα μας ξεπεράσουν οι Αμερικανοί γιατί ακριβώς το ίδιο ε, κάνουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χολμαϊερ.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 έχει θέσει πέντε μετρήσιμους στόχους για την Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 που επικυρώθηκαν από τις χώρες μέλη και μας δίνουν μια κατεύθυνση. Η επιτυχία, της, επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από το πώς θα τους αφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρτάται επίσης από την υπευθυνότητα που θα επιδείξουν οι διάφορες χώρες μέλη, αν θα καταφέρουν να αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης, να περιορίσουν την εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά πριν ε, το τέλος της σχολικής ηλικίας, αν θα μειώσουν τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην ένδια και αν θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, κλιματικές αλλαγές. Παρόλο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συμφωνία, η χώρα μου αποφάσισε να περικόψει διάφορα τέτοια προγράμματα και τα χρήματα θέλει να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει δρόμους μετά από διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, εσείς ε, προσωπικά αλλά και συλλογικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζετε την ε, θέση αυτή να πάμε προς μια κατεύθυνση η οποία δεν είναι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μπένοβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο προπολογισμό είναι ένα στοιχείο κλειδί βέβαια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πολλά εξαρτώνται από τον προπολογισμό. Σε περίοδο κρίση, ο κοινοτικό προπολογισμό μπορεί να συνεισφέρει, να απαλύνει κάπω την πολιτική λιτότητα που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη-μέλη και να βάλει χρήματα σε επενδυτικά προγράμματα. Η έκθεση αυτή υποστηρίζει δαπάνες και στις υποδομές. Δεν θα πρέπει όμως να αποτελούν αυτά τα, συγγνώμη, αυτά ομόλογα, τα διευθυντικά, να αποτελούν υποκατάστατο των ευρωομολόγων. Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν συμφωνώ με την ιδέα περιορισμού του κοινοτικού προπολογισμού. Δεν βοηθά την ολοκλήρωση, ούτε την οικονομία, ούτε και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Οι εγωισμοί θα πρέπει να πάψουν να χωρίζουν την Ευρώπη σε αυτούς που πληρώνουν και σε αυτούς που πληρώνονται. Η αλληλεγγύη, αυτό είναι το σημαντικό στην Ευρώπη και αυτό βοηθά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο, οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2012 θα επηρεάσουν το μέλλον. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε οικονομίες τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το μηνιαίο ε, έξοδο που κάνουμε για να πηγαίνουμε από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο κάτι που εκνευρίζει τους πολίτες μας, τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Το 2012 λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε και να κοιτάξουμε αν υπάρχει δυνατότητα να μειώσουμε τα ταξίδια αυτά ή τέλο πάντων να αλλάξουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Ένα άλλο θέμα είναι το Ευρωπαϊκό Μουσείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αναβληθεί τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, να περιμένουμε μια καλύτερη στιγμή για την Ευρώπη. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να δαπανάμε χρήματα για το 2012, αντίθετα να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και δουλεύουμε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σμόλκοβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, η οποία ονομάζει τα πράγματα με το όνομά τους. Ο προπολογισμό 2012 και μετά πρέπει να είναι φιλόδοξο, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να πετύχουμε του στόχου τη στρατηγική μα για το 2020 μετά την κρίση και να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο. Η ιδέα ε, συνάντηση Επιτροπή Προπολογισμών με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι καλή. Μπορούμε έτσι να συζητήσουμε και τους προϋπολογισμούς τους εθνικούς για το 2012. Ο κοινοτικό προπολογισμό μπορεί να μην είναι ελληματικό, είναι 2% των ε, δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στου εθνικού προπολογισμού και τον κοινοτικό προπολογισμό. Ο κοινοτικό προπολογισμό σχεδιάζεται για να επενδύσει στο μέλλον τη Ευρώπη. Το Συμβούλιο πρέπει να το κατανοήσει αυτό. Έχουμε ήδη εκπροσώπου από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που θέλουν να παγώσει ο κοινοτικό προπολογισμό, κάτι το οποίο θα επιβραδύνει την ανάπτυξη τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε, ο Επίτροπο Λεβαντόσκι έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε. Πρόεδρε, τρία σημεία μόνο. Στρατηγική 2020 και την προσαρμογή της ε, κυρία Μπαλσάνη με την πρότασή τη. Το 41% των δαπατών, των δαπανών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προβλέπονται για το στόχο του 2020. Το ίδιο γίνεται και με την ε, προβλησμό του 2012. Αλλά προσπαθούμε εμείς να προσαρμόσουμε το πλαίσιο. Μέσα στα πλαίσια βέβαια του προπορισμού 2007-2013. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες ε, ελιγμού που έχουμε και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να κινηθούμε. Βέβαια τώρα για αυτό που είπε ο κύριος Έλλης, αλλά και ο κύριος Γκάιερ και η κυρία Ολμάιερ, όσον αφορά τις ανητικές ε, προτεραιότητες, φοβούμε, και αυτή είναι η πραγματική ιστορία για το προπορισμό του 2012, ότι σήμερα ε, ε, πρέπει να, εκτός από τις θετικές προτεραιότητες, να δούμε και τι δεν λειτουργεί τι δεν ε, την χάνει σωστούς, ε, σωστές διαχειρίσεις για να κάνουμε και εξοικονομήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει ο προβλησμός να ασχοληθεί και με θετικές αλλά και αρνητικές προτεραιότητες. Όσον αφορά την αυστηρή διαχείριση, αυτό είναι πραγματικά μία αναγκαιότητα. Ε, βέβαια το θέμα της διαχείρισης και της διοίκησης είναι 4,7% του σφαιτικού προπολογισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι γνωστή η Ολλανδία για πολύ συνετή προσέγγιση στις δαπάνες. Ο προλογισμός μας δεν έχει έλλειμμα και δεν μπορεί να θεωρηθεί να κατηγορηθεί ότι σπαταλά τα χρήματα όπως γίνεται σε πολλά κράματα. Το σκεπτικό το παρουσίασε ο κύριος Γεμπράντη όσον αφορά την οριμότητα των προγμάτων και όσον αφορά την αξιοπιστία. Γιατί εδώ έχουμε πραγματικά τις δεσμεύσεις για τις πληρωμές και σε περιόδους λιτότητας πρέπει κανένας να πληρώνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα ε, αξιοπιστίας, είναι θέμα συνοχής, είναι θέμα ε, επένδυσης κατά κάποιον τρόπο των χρημάτων. Και αυτό νομίζω ότι απαντά σε εκείνους που βρίσκεται τώρα εκτός του Κοινοβουλίου και ε, κάνουν μια διαδήλωση. Ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε κυρία Βαλζάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τις ε, τοποθετήσεις ακούστηκε πολλές φορές η λέξη ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας, ούτως ώστε οι πολίτες να μην μείνουν μόνο με τα λόγια μας. Πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτά που κάνουμε και που λέμε τα μεγάλα σχέδια είναι η στρατηγική του 2020. Πρώτος στόχος είναι περισσότερη δουλειά, δεν είναι μόνο φιλόδοξο. Είναι συγκεκριμένο, έχουμε, το μετράμε με τις παραμέτρους μείωσης της ανεργίας. Πρόκειται για έναν ειδικό και πολύ φιλόδοξο στόχο και θεωρώ εγώ ότι είναι θεμελιώδες να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν τον στόχο, γύρω από αυτόν τον στόχο για να τον προσεγγίσουμε. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ φιλόδοξη η στρατηγική του 2020 για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα και μόνο έγγραφο τον προϋπολογισμό, τότε θα αποτύχουμε. Και υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Η λιτότητα δεν είναι πολιτική, δεν είναι μέσο, είναι ένας όρος για τον εναντίον του οποίου πρέπει να αντιδράσουμε όχι μόνο ενισχύ, σταθεροποιώντας τη δαπάνη αλλά με διαφορετικά μέσα από αυτά των εθνικών προϋπολογισμών. Διαφορετικό μέσο σαν αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να κάνουμε κάτι το καινούργιο φέτος. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Χρειάζεται να ορίσουμε μια νέα στρατηγική, να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και των δικών μας προϋπολογισμών προπολογισμού. Πρόκειται για ένα μέσο απόλυτα ευρωπαϊκό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους όρους πραγματοποίησης της στρατηγικής 2020. Ολοκληρώνουμε την συζήτηση, διακόπτουμε μέχρι τις 11.30 την Ολομέλεια, όπου θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία.